Απαγόρευση δηλαδή τεχνολογιών που χρησιμοποιούν και ανούχα άλατα για την εξόριξη μετάλλων. Εδώ έχουμε τον κύριο Μεσάρος που θέλει να κάνει επεξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να επεκταθεί η απαγόρευση χρήσης και ανιούχων ουσιών στην εξόρυξη στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταργηθεί τελείως, να καταληφθεί τελείως αυτή η τεχνολογία για να αποφευθούν και περαιτέρω σοβαρές ε, φυσικές ε, θεομηνίες ε, τοξικά απόπλητα που καταλήγουν στον υδροφόρο ορίζοντα. Έχει εξαφανιστεί, έχει εξολοκληρωθεί όλη η πανίδα του ποταμού Τίσα στην Ουγγαρία και στη Σλοβακία επίσης γιατί συνέβη ένα ατύχημα κοντά στα σύνορα. Να μην ανοίγουν τέτοια ε, ορυχεία με χρήση ε, τέτοιων ε, επικινδύνων τεχνολογιών. Και δεν είναι καθόλου διμερές θέμα κρατών μελών. Είναι προς κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι η πολιτική μας βιώσιμη. Γι' αυτό υπερψήφισα την έκθεση και θα ήθελα να ενώσω και εγώ τη φωνή μου με όσοι υποστηρίζουν τα μέτρα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμείς είμαστε υπέρ της απαγόρευσης χρήσης εξόριξης ε, ε, μάλλον, υπέρ της απαγόρευσης της χρήσης και ανιούχων ε, ε, αλάτων στην εξόρυξη μετάλλων και προκαλούν τεράστιους κινδύνους στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Με την ψήφο μας θελήσαμε να εκφράσουμε τη σαφή μας βούληση ω ως αντιπροσωπεία, Ιταλική αντιπροσωπεία του Άλτε να μην διαπραγματευτούμε θεμελιώδη δικαιώματα όπως η υγεία των ανθρώπων και η διατήρηση της φύσης για χάρη λίγων ε, ε, λίγων εγκαταστάσεων και εφόσον πρόκειται για εξόριξη χρυσού και σίγουρα όχι για πατάτες αυτοί, αυτές οι εταιρείε θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του που είναι απαραίτητοι για την έρευνα και για την τεχνολογία που να είναι συμβατή με το περιβάλλον και με την προστασία της υγείας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Ουγγίας. Ο κύριος Βατίμ Τούντορ. Ευχαριστώ ε, κυρίες και κύριοι. 500 συνάδελφοι εχθές ε, ψήφισαν συντριπτικά κατά της χρήσης ε, των κιανιούχων στα ορυχεία. Γίνεται λόγος για το κιάνιο. Όταν λέμε κιάνιο εννοούμε θάνατο και αφορά και εμάς τους Ρουμάνους. Έχουμε από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού παγκοσμίω και ουράνιο. 300 ε, τόνοι ε, ουράνιο, ε, ασίμι, χρυσό, σπάνιες γέες. Έχουμε πάρα πολλά ορυκτά στη Ρουμανία. Δεν μπορούν οι πολυεθνικές να χρησιμοποιούν τέτοιες επιθετικές μεθόδους και μετέρχονται και κάθε μέσου και γελία ψέματα χρησιμοποιούν. Κάνουν όμως τεράστια καταστροφή θέλουν να καταστρέψουν με δυναμίτη τέσσερις λόφους, εννέα κημητήρια και ε, διάφορες εκκλησίες χριστιανικές. Χιλιόμετρα ε, ολόκληρα ε, ορυχείων θέλουν να καταστρέψουν παλιές τοές που είναι μοναδική κληρονομιά μέχρι και η UNESCO το έχει αναγνωρίσει. Έχει ζήσει ένα Τσερνομπίλ Ευρώπη. Δεν χρειαζόμαστε και δεύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Μπρέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα χθε κατά του ψηφίσματος διότι αυτό μου ζήτησε η τοπική κοινότητα. Οι τοπικές κοινότητες εκεί θεωρούν το ψήφισμα αυτό, θεωρούν ότι αντιβαίνει στην ανάπτυξή τους. Ζητήθηκε από ορισμένου συναδέλφου μελέτη που θα διευκρινίσει τι συνέπειε, τι επιπτώσει στο περιβάλλον. Μια τέτοια ενέργεια είναι ορθή. Αλλιώ τα πάθη που έχουν αναμειχθεί πλέον στη συζήτηση αυτή δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να καταστρέψουν οποιασδήποτε πιθανότητε έχει να αναπτυχθεί η κοινότητα αυτή στο μέλλον. Σα ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με την πρώτη έκθεση Μέντε Τεβίγο. Η κυρία Οβίρ. she not. από ό,τι φαίνεται η κυρία Οβίρ δεν είναι παρούσα. Ακολουθεί η έκθεση, δηλαδή επεξηγήση ψήφου για την έκθεση για το Κυργιζιστάν. Πρώτα ο κύριος Higgins. Νομίζω τον βλέπω να σπέβδει προς το μικρόφωνο. And you have the floor, Mr. Higgins. Yes, uh, thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, γιατί επιτρέπεται τόσο ανεδός να μιλούν μεγαλόφωνα οι συνάδελφοί μου ώστε να μην μπορεί κανείς να λάβει το λόγο. Ο πρόεδρος. Μας μένουν 5 με 10 λεπτά πριν να έλθει εδώ ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, κ. Biden. Σας παρακαλώ λοιπόν κάντε κάποια ησυχία για να μπορέσουν να μιλήσουν να μιλήσουν σε αξιοπρεπέ περιβάλλον οι συνάδελφοί μα. Ο κ. Higgins. Απέσχον ε, στο ψήφισμα για το Κυρκυζιστάν. Προπενταετίας ο λαός του Κυρκυζιστάν κινητοποιήθηκε ενώ την επανάσταση της ε, Τουλίπας για να ρίξει το διεφθαρμένο καθεστώς και να βελτιώσει τη ζωή του. Δυστυχώς η εξουσία που ακολούθησε κατεπρόδωσε τις ε, προσδοκίες των μαζών καθιδρύοντας νέο διεφθαρμένο καθεστώς. Δεν πιστεύει ο κόσμος πλέον ότι θα βελτιωθεί η ζωή του. Εγώ υποστηρίζω τους φίλους μου σοσιαλιστές από την Αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή που ζήτησε να γίνουν εκλογές για νέο κοινοβούλιο και που κατέστησε σαφές ότι δεν πρόκειται τίποτε να αλλάξει αν δεν προβληθούν νέοι υποψήφοι από τις ε, μάζες που, που ζουν στην Ήπεθρο αλλά και στις πόλεις. Για να αντιμετωπίσει την καταστροφή που έχει προκύψει τα τελευταία 20-25 χρόνια, να αντιμετωπίσει τον νέο καπιταλισμό, να φέρει πραγματική νέα δημοκρατική πνοή με θεσμούς που θα βασίζονται στην κοινή εκφρασμένη βούληση των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ. έκθεση Πέτερλε, η ε, κυρία Μικουλιένε. Παρακαλώ ησυχία. Ευχαριστώ. Το κείμενο αυτό αγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία, χωρίς αντίδραση. Και βεβαίω είναι κατανοητό αυτό, διότι μα ενδιαφέρει και μα αφορά όλου η δημόσια υγεία. Συγχαίρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλου του Ευρωπαίου πολίτε, καθώ επίση και την εισηγητή του Κοινοβουλίου για την πρόταση αυτή και θα ακολουθήσουν και άλλα έργα και άλλες πράξεις για την καταπολέμηση του καρκίνου και για να λάβουμε και προληπτικά μέτρα κατά του καρκίνου, διότι η κατάσταση σήμερα είναι ανησυχητική. Θα πρέπει να ε, κινητοποιηθούμε για να λύσουμε τα προβλήματα αυτά. Είμαι πεπισμένη ότι η καθολική προσέγγιση πλήρης ε, απέναντι στο καρκίνο θα πρέπει να είναι προτεραιότητα και εθνική μας και ευρωπαϊκή. Θα πρέπει να ε, ενταχθεί στη στρατηγική μας για τη δημόσια υγεία να έχουμε συντονισμένες ενέργειες για να μειωθεί ο καρκίνος. ευχαριστώ. Ο κύριος Πάσκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έκθεση για την καταπολέμηση ε, του καρκίνου είναι ε, κάτι που πρέπει να τονιστεί και να τονιστεί ακόμα περισσότερο η σημασία της πρόληψης σε περίπτωση έγκαιρης διάγνωσης γνωρίζουμε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες πλήρους θεραπείας. Υπάρχουν κάποιες ε, ε, προδιαθέσεις κληρονομικές ή ο τρόπος ζωής που ευνοούν την ε, ανάπτυξη καρκίνου. Είναι καλός λοιπόν ο προσυμπτωματικός έλεγχος, το screening, για να προλαμβάνει το καρκίνο. Το επόμενο βήμα θα μπορούσε να είναι να επεκταθούν, να διευρυνθούν όλες οι θεραπείες σε όλα τα κράτη-μέλη και σε μικρές κλινικές, όχι μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία και σε μέρη που δεν υπάρχει μεγάλη εμπειρία για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιβίωσης. Εν πάση περιπτώσει, ε, τιμώ τον κύριο Πέτερλε και ε, την έκθεσή του και ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε τον καρκίνο όπω χρειάζεται στην Ένωση. Ευχαριστώ κύριο Μπονσινιόρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την ε, Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων και θα ήθελα όλος ιδιαίτερος να ε, συγχαρώ τον εισηγητή, τον κύριο Πέτερλε. Έχει κάνει μια πρόταση πάρα πολύ καλή ε, συνεργασίας για την καταπολέμηση του καρκίνου είναι, ξέρετε, ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο για όλους μας και λεπτό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, 2 εκατομμύρια Ευρωπαίων χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους από καρκίνο. Και 10% των ε, περιστατικών αυτών οφείλεται στην έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες στον χώρο εργασίας θα πρέπει να μειωθούν αυτά τα κρούσματα κατά 15% μέχρι το 2020. Είναι ένα στόχος πάρα πολύ αξιόλογο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποδείξει την ενότητά της και ε, στα πλαίσια της συγκεκριμένη δράση Και το άρθρο 66 είναι πάρα πολύ σημαντικό προ την κατεύθυνση αυτή. Πρόκειται γιατί διάθεση των φαρμάκων σε όλους και σε όλες τις χώρες. Γι' αυτό υπερψήφισα εγώ και την έκθεση. Ο Πρόεδρος, ξέρω ότι είστε πολύ ανυπόμονοι και δημονείτε να δείτε τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά 5 με 10 λεπτά ακόμα θα καθυστερήσει, οπότε προσπαθήστε να είστε λίγο ήρεμοι για να ακούμε τους συναδέλφους. Επόμενη έκθεση, επεξήγηση ψήφου, η έκθεση της κυρίας Τόγια, κινητοποίηση των τεχνολογιών, προφοριών και επικοινωνιών. Ο κύριο Μεσάρο θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η τεχνολογία των πληροφοριών και των επικοινωνιών έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Ο κλάδος συνεισέφερε με την ανάπτυξή του ε, στην εξέλιξη και στην ανάπτυξη και άλλων ε, κλάδων της τεχνολογίας ε, που είναι η τεχνολογία των μετρήσεων και η νανοτεχνολογία και είχαν αποτελματωθεί. Γι' αυτό εμείς καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χρησιμοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες για να πληρώσει τους στόχους για το 2020. Χαίρομαι που είχα την ευκαιρία να υπερψηφίσω την πρωτοβουλία αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό μέχρι το 2020 να έχουμε καλύψει τους στόχους μας και να έχουμε τεχνολογίες αποτελεσματικές και αποδοτικές που να εξοικονομούν ενέργεια. Είναι στρατηγική σημασία ο κλάδος αυτός των επικοινωνιών και των πληροφοριών για να φτάσουμε στους στόχους μας. Γι' αυτό χρειάζεται όμως τυποποίηση ε, των ε, μηχανημάτων και συσκευών μέτρησης και ένα πακέτο πρωτοβολιών που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη για των υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Επόμενη έκθεση, έκθεση πρώτη. Τρεις ομιλητές έχω. Η κυρία Ματέρα πρώτη. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι υπέρ και στηρίζω την ε, πολύ αξιόλογη δουλειά του συναδέλφου Βιτόριο Πρόντι που αποτελεί την, ε, την αίσια κατάληξη που, είχε η πρόταση της Ελλάδας. Εγώ εκπροσωπώ το νότο της Ιταλίας που βρέχεται από την ε, λεκάνη της Μεσογείου. Έτσι έχουμε εμπιστοσύνη πως δεν θα είμαστε απροπαϊκοί ετοίμαστε έναντι των ε, επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στις περιοχές μας που ζουν ε, βασικά από τη γεωργία, την αλληλεία και τον τουρισμό και που είναι σε μεγάλο βαθμό, που αποτελούνται από σε μεγάλο βαθμό από κοινότητε και κοινωνικές ομάδες πιο αδύναμες, πιο ευάλωτες. Θεωρώ πως είναι σε μελιώδες η αλληλεγγύη ανάμεσα στη ε, κράτη και στις διαφορετικές περιφέρειες και η απάντηση με αυτή τη νέα στρατηγική που τώρα φτιάχνουμε είναι πολύ ικανοποιητική. Φυσικά με όλη αυτό το θόρυβο είναι πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς. Ωστόσο είμαι υπέρ αυτού του, του, της έκθεσης αλλά και να σας θυμίσω το μηχανισμό αλληλεγγύης που θα λειτουργήσει για σύντομη, για, γρήγορα για περιπτώσεις ε, κλιματικών αλλαγών. Πραγματικά είναι αδύνατο να μιλήσει κανείς εδώ μέσα. Κυρία Αντρικένε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Υποστηρίζω το λευκό βιβλίο της Κομισιόν και την έκθεση του κ. Πρόντι. Νομίζω πως αυτό το λευκό βιβλίο χρειάζεται μετά από το, οι διαπραγματεύσει Κοπεχάγη για τι κλιματικέ αλλαγέ. Ε, δεν είναι αρκετά τα όσα αποφασίστηκαν εκεί. Το μη δεσμευτικό έγγραφο που συμφωνήθηκε στην Κοπεχάγη για να σταματήσει η παγκόσμια ε, υπερθέρμανση του πλανήτη θα σημαίνει και πάλι ε, προσπά... μεγάλες προσπάθειες ε, για την Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάζεται να προσέξουμε ιδιαίτερα τον τρόπο με τον οποίο προπαράγουμε ενέργεια. Πρέπει να καταβάλουμε ε, εντονότερες προσπάθειες για να, ε, όσον αφορά την ενεργειακή μας πολιτική, αλλά και να προωθήσουμε την έρευνα σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. αλλά και να εξετάσουμε πώς οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να ενταχθούν στο ενεργειακό μας ε, μείγμα. Ευχαριστώ. Frau Kadenbach, bitte. Ευχαριστώ κυρία Κάλενμπαχ, παρακαλώ. Ναι, υποστηρίζω και εγώ την ε, αίτηση του κυρίου Πρόεδρη. Αυτό όμως ε, που με προβληματίζει είναι μια τροπολογία που ενέκρινε η Ολομέλεια για την έκθεση αυτή ε, που ήταν η τροπολογία του κυρίου Σέμπερ και του Λαϊκού Κόμματος. Φοβούμαι ότι με αυτόν τον τρόπο οι συντηρητικοί θα μας βάλουν από το παραθυράκι και πάλι την πυρηνική ενέργεια. εκθιάζεται ε, η πηγή ε, αυτή η ενέργειας που δεν ε, παράγει διοξίδια του άνθρακα. Αυτό είναι παλιά πάγια τακτική του λόμπι της πυρηνικής ενέργειας. Και εγώ ως Αυστριακή δεν καταλαβαίνω. Δεν την, δεν την αντιλαμβάνομαι ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας στην πυρηνική ενέργεια. Και δεν μου αρέσει καθόλου. Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε αυτή την παράγραφο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Λοιπόν, Αγαπητοί συνάδελφοι, διακόπτονται οι επεξηγήσεις ψήφου και ακολουθεί η πανηγυρική συνεδρίαση.